Ωραία. Τα πρακτικά θα διανεμηθούν στην επόμενη σύνοδο και αν δεν διαφωνεί κανείς θα θεωρήσω εγκεκριμένα τα ψηφίσματα. Μάλλον θα τα διαβιβάσω αρμοδίως τα όσα εγκρίναμε.